συνεισφέρατε σε αυτή την εξαιρετική συζήτηση. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά ε, θα δώσω τη σκητάλη στην φίλη και συνάδελφο την κυρία Καϊλή έτσι θα μπορέσω να παρακολουθήσω και εγώ τη συζήτηση χωρίς να εργάζομαι, που ασχολείται με την, είναι επικεφαλής μάλλον της Επιτροπής ΣΤΟΑ. Συμμετείχα στην Επιτροπή αυτή που κάνει πολύ καλή δουλειά και πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κυρία Καηλή και σας παραδίδω τη για να προεδρεύσετε στο επόμενο πάνελ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Θα μας λείψετε κυρία Αντιπρόεδρε. Έχω δουλέψει σε πολλούς φακέλους όπου παρακολουθώ τι συμβαίνει με τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται, το μέλλον ε, υπάρχει αυτό το πάνελ για το μέλλον και την τεχνολογία. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζουμε πώς ε, έχουν αντίκτυπο στην ζωή μας αυτές τι τεχνολογίες, πώς ε, αλλάζουν τη ζωή μας και βεβαίω πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμεί σε νομοθετικό επίπεδο. Πριν από τρία χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη αντιληφθήκαμε ότι αλλάζει τα πάντα αλλάζει όλους τους τομείς της ε, καθημερινότητάς μας. Αρχίσαμε λοιπόν να ζητούμε νομοθεσία πριν από τρία χρόνια και να, και να ζητάμε και έναν ηθικό κώδικα, ένα κώδικα ηθικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε κάνει πολλή δουλειά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και χαίρομαι που γίνεται αυτή η ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους ε, θρησκειών, εκκλησιών αλλά και φιλοσοφικών οργανώσεων η ηθική ήταν πάντα προτεραιότητά μας και αντιλαμβανόμαστε ότι θα αποτελέσουμε μια σημαντική πρόκληση. Επίσης η ΣΤΟΑ συνεισέφερε με τρία έγγραφα ενημέρωσης, briefing που πρέπει να έχετε λάβει και μπορεί να δείτε τι δουλειά έχουμε κάνει εμείς έως τώρα και βεβαίω μας περιμένουν και άλλη δουλειά και, άλλη, και άλλα τέτοια έγγραφα. Προσπαθούμε να εξετάσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης ε, στην υπηρεσία της κοινωνίας, ε, στην υπηρεσία του καλού δηλαδή, αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ της πτυχής ε, της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητονεμοσύνη και των Πολιτειών ή της Κίνας. Για μας η βασική προτεραιότητα είναι πως αυτό θα είναι υποφελής για τους πολίτες, όχι μόνο πως θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί παγκοσμίω. Βεβαίως υπάρχει και αυτή η πρόκληση, όμως πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τους πολίτες μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον καθηγητή Τόμας Μέτσιγκερ, που είναι μέλος της, της ομάδας υψηλού επίπεδου για την ε, τεχνητή νοημοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, έχουν προετοιμάσει οι κρατικές γραμμές για την ηθική τεχνητή, τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω πως παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτό. Ακούσαμε, ε, έτσι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ε, είναι και η Ashley Fox εδώ που είναι που είναι μάλλον ε, εισηγητή ε, για την τεχνητή νοημοσύνη και συνεργαστήκαμε στον τελευταίο σημαντικό φάκελο πριν το τέλο τη θητεία μα. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσε ιδέε που μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτό το φάκελο. Υπήρξε μεγάλη υποστήριξη για το ε, κείμενο αυτό. το αναφερθώ σε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία αυτού του κειμένου. Το, το μέσο τη κοινωνική και ηθική ευθύνη, τεχνητή νοημοσύνη, θέλουμε να υπάρχει η ηθική να, να περιλαμβάνεται ήδη στον αρχικό σχεδιασμό, ethics by design και βεβαίω πρέπει να υπάρχουν κυρώσει όταν υπάρχει χειραγώγηση τη αντίληψη τη τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε, έρχονται και εκλογέ και θα μπορούσε ε, κάποια κόμματα, θα μπορούσαν κάποια κόμματα να ευνοηθούν ε, κάποια βίντεο με βίαιο περιεχόμενο οδηγούν παραδείγματος χάρη σε πιο συντηρητικές απόψεις ή το αντίθετο ε, πρέπει οπωσδήποτε οι διακρίσεις να μην έχουν θέση στην Ευρώπη στην, ε, στο ζήτημα αυτό. Το βλέπουμε αυτό σε πολλές πλατφόρμες. Όταν υπάρχουν διακρίσεις ε, χρειαζόμαστε κανόνες γι' αυτό για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Επίσης ζητάμε και κέντρα αριστεία στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση Θέλουμε δηλαδή να αναπτύξουμε τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια για να προστατευτούμε από όλα αυτά. Επίσημη λοιπόν ε, ε, υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη με ηθικές αξίες και αρχές θα έχουμε και προσώπους ε, από την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Καθολική Εκκλησία, από τον, την ανθρωπιστική κοινότητα. Όλοι αυτοί οι φορείς έχουν παράδοση ε, σκέψης και συνεισφοράς ε, σε ό,τι φορά ε, την, την ανθρωπότητα και το μέλλον της. Αν δεν υπάρχει χώρος για σας εδώ μάλιστα. Εντάξει, θα δώσω, σας δώσω το λόγο τώρα ως πρώτος ομιλητής. Κύριε Μέτσιγκερ, έχετε το λόγο. Α, σας βλέπω τώρα. Θέλω να σας πω ότι είμαι κουρασμένος, εξαντλημένος. Έρχομαι εδώ από μια συνάντηση της ομάδας υψηλού επίπεδου για την ε, ε, τεχνητή νομοσύνη. Τις τελευταίες δύο ημέρες δουλέψαμε πολύ σκληρά ε, και το, η καλή είδηση είναι ότι έχουμε φτάσει ε, φτάσαμε σήμερα στο τέλος ε, τη σύνταξη αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών. Ε, θα σας τα δώσουμε σήμερα ή αύριο. Πάντως, με πάση περιπτώσει, την Παρασκευή θα έχετε την τελική εκδοχή του εγγράφου, το οποίο θα δημοσιευτεί στις 8 Απριλίου μπορείτε όλοι να είστε σίγουροι ότι όταν το διαβάσετε το έγγραφο αυτό θα νιώσετε έτσι μια ανάταση, ένα αίσθημα πολυθετικό και όταν όμως θα διαβάσετε το έγγραφο για δεύτερη φορά θα διαπιστώσετε ξαφνικά ότι σε αυτό υπάρχουν ε, κενά, ελλείψεις ε, και δεν υπάρχουν έτσι κανονιστικές ρυθμίσεις σε αυτό το έγγραφο. Θα δείτε όμως ε, στην αρχή ότι θα εντυπωσιαστείτε και θα σας αρέσει το έγγραφο. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Δηλαδή το πώς ακριβώς ε, συντέθη αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου. Η δική μας δουλειά ήταν να καταλήξουμε στις κατευθυντής γραμμές ηθικής για την Ευρώπη. Αλλά από τα 52 μέλη είχαμε μόνο τέσσερις φιλοσόφους, τέσσερις ε, που ε, στην προηγούμενη ζωή τους είχαν μια εκπαίδευση στην ηθική. Και βλέπετε ότι υπήρχε ουσιαστική εκπροσώπηση των ε, βιομηχανικών κύκλων στην ομάδα, θα το δείτε αυτό ότι ε, έχει παρισφρήσει και στο κείμενο. Έμαθα ε, πολλά πράγματα τους τελευταίους εννέα μήνες που δούλεψε σε αυτή την ομάδα. Πολύ έξυπνοι και πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι. Ένα πράγμα που όλοι πρέπει να ξέρετε είναι το περίφημο ethics washing. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει να καλλιεργούμε ηθικές συζητήσεις γιατί θέλουμε να καθυστερήσουμε, να αναβάλουμε, να αποφύγουμε ή να αποτρέψουμε ανθρώπους ε, από ε, το να εκπονήσουν κανόνες για την πολιτική. Αυτό είναι ο βασικός ε, στόχος της βιομηχανίας, δηλαδή να μην υπάρχουν νόμοι που να εφαρμόζονται. Παραδείγματο χάρη, το Facebook και η Amazon. Αυτό ε, τους αρέσει να έχουμε έτσι μακρές ηθικές συζητήσεις στην Ευρώπη, γιατί όσο πιο πολύ διαρκούν αυτές οι συζητήσεις, τόσο περισσότερο χρόνο ε, έχουν και αυτοί πριν αρχίσουν να ισχύουν οι νόμοι. Επίσης, χρειαζόμαστε νόμους που να είναι δεσμευτικοί ε, και να έχουν νομιμοποιηθεί από δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν πρόκειται μόνο για την ηθική. Αν δούμε λοιπόν πώς ακριβώς περιγράφουμε τους εαυτούς εαυτούς μας. Ένα από τα βασικά σλόγγαν είναι η ηθική ως μια αναγκαιότητα ε, που θα δώσει τη δυνατότητα να γίνονται δουλειές, ε, δουλειές με δέλτα κεφαλαίο και έτσι λοιπόν ε, αποκτάτε και εσείς μια ιδέα για τη στρατηγική που βρίσκεται πίσω από αυτό το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στις 8 Απριλίου. Για ορισμένους ανθρώπους αυτό είναι μια δήλωση για στρατηγικές επενδύσεις. Ακούσαμε ήδη την έννοια του shopping, ε, του να αγοράζει κανείς ηθική. Και ο κίνδυνος είναι ότι αν υπάρχουν άκαμπτοι κανονισμοί στην Ευρώπη, η έρευνα θα μετακινηθεί σε άλλα μέρη του κόσμου. Όμως ε, Βλέπουμε ότι το Facebook ήδη αντιδρά, αγόρασε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο όπου θα εκπαιδεύει τους δικούς της τους ε, αρμόδους για ηθική. και αυτοί ε, θα μπουν στην Ευρώπη γιατί και οι βιομηχανικοί κλάδοι δημιουργούν ε, τη δική τους ηθική, τουλάχιστον στην πατρίδα μου. Θα ήθελα να σας αναφέρω και ένα παράδειγμα ε, πριν σιγά σιγά περάσω και στο θέμα της σημερινή μας συνάντησης. Ε, μου ανετέθη να εισηγηθώ τις κόκκινες γραμμές για την Ευρώπη. Οι κόκκινες γραμμές είναι αδιαπραγμάτευτες ηθικές αρχές. Πράγματα τα οποία ε, δεν θα θέλαμε ποτέ στην Ευρώπη υπό καμία προϋπόθεση. Δουλέψαμε για πολλούς μήνες με πολλούς εμπειρογνώμονες ε, και όταν λοιπόν καταλήξαμε σε έναν κατάλογο κόκκινων γραμμών η βιομηχανία είπε η λέξη κόκκινη γραμμή δεν μπορεί πια να υπάρχει μέσα σε αυτό το έγγραφο σε κανένα σημείο. Η βιομηχανία, η βιομηχανική κύκλοι είπαν ότι η λέξη αδιαπραγμάτευτος ε, πρέπει να αφαιρεθεί από το έγγραφο. Στο έγγραφο του, της 8ης ε, Απριλίου θα διαβάσετε ότι τίποτα δεν είναι πια διαπραγμάτευτο, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι οτιδήποτε μπορεί να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση. Παζάρι δηλαδή στο μέλλον, όπου δεν θα υπάρχουν αποδεκτές ηθικές ε, γραμμές, αλλά η βιομηχανία θέλει ε, να προβεί σε αυτήν την διαπραγμάτευση. Και η δυσάρεστη είδηση για το έγγραφο αυτό είναι ότι οι ηθικές κατευθυντήριες γραμμές θα δημοσιευτούν, αλλά θα έχουν το βασικό, το κεντρικό αποτύπωμα της βιομηχανίας. Γίνεται λόγος για την νομική δομή, αφηρημένα στοιχεία, πολλά ανεπίλητα θέματα. Πρέπει να σου χάνει το θέμα του ε, πώς μπορούν να εξηγηθούν πολλά. Ε, αυτό συγκαλύφθηκε θέματα όπως η τεχνητή συνείδηση ή η τεχνητή γενική νοημοσύνη. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά και πάρα πολλά ερωτήματα των Ευρωπαίων πολιτών που δεν έχουμε απαντήσει και το έγγραφο αυτό ε, είναι κοντόφθαλμο. Δηλαδή δεν εξετάζει το μακροπρόθεσμο ή έστω μεσοπρόθεσμο μέλλον. Βέβαια υπάρχουν και ε, ευχάριστες ειδήσει ότι αυτή τη στιγμή οι κατευθυντήριες γραμμές ηθικής είναι πολύ καλύτερες από οτιδήποτε έχουν η Κίνα ή οι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχω δει πολλές από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και ευχαριστες ειδησει οτι αυτη τη στιγμη οι κατευθυντηριες γραμμες ηθικη ειναι πολυ καλυτερες απο οτιδηποτε εχουν η κινα η οι ηνωμενε πολιτειε εχω δει πολλε απο αυτες τι κατευθυντηριε γραμμε και θελω να σα πω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχουμε εμείς. Άρα δηλαδή είναι ένα θαυμάσιο πρώτο βήμα για να ακολουθήσει ένα δεύτερο, δηλαδή μια πλατφόρμα για συζήτηση. Και τι χρειαζόμαστε τώρα, κατά την άποψή μου, χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Μια νέα γενιά εμπειρογνωμόνων ε, στην ε, ηθική της τεχνητής γνωμοσύνης. Χρειαζόμαστε περισσότερη επαγγελματική έρευνα, να συνεχιστούν οι συζητήσεις ε, με λιγότερες προκαταλήψεις Χρειαζόμαστε συζητήσεις, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Χρειαζόμαστε τη διάδοση των ε, ερευνητικών πορισμάτων στο κοινό ε, και επίσης και στους ε, φοιτητές. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας και τους φοιτητές για όλα αυτά. Μία λοιπόν θετική πρόταση είναι το το 12% των επενδύσεων που θα είναι 20 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος κατά τα επόμενα έτη να τα ε, διοχετεύσουμε σε ένα κέντρο για την ηθική και σε ένα εκπαιδευτικό δίκτυο σε όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και σε όλες τις χώρες. Προτείνω λοιπόν να συνεχίσουμε τη συζήτηση που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στην ομάδα υψηλού να περάσει το όλο θέμα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όλα τα πανεπιστήμια και να σας ενημερώσω ότι το MIT το έχει ήδη κάνει. Μόλις επένδυσε ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να υπάρχει ένα κέντρο για την τεχνητή νοημοσύνη. Και τώρα ένα μεγάλο ερώτημα που θέτω σε όλους εσάς είναι σε αυτήν την κρίσιμη ιστορική μετάβαση ε, η συμφωλή των ανθρώπων, η ανθρωπιστική, η θρησκευτική, ε, ποια μπορεί να είναι με βάση όμως ουσιαστική συνεισφορά, με βάση επιχειρήματα. Καθόμουν εκεί στη γωνία και άκουσα ε, τα πρώτα 90 λεπτά και παρακολούθησα πολλούς νέους που έφυγαν και θα διαπιστώσετε ότι η αίθουσα είναι λίγο πιο άδεια από τότε που ξεκινήσαμε. Και ίσως ε, να το γνωρίζετε αυτό, Υπάρχει ανταγωνισμός. Θα γνωρίζετε ίσως ότι υπάρχει μια νέα θρησκεία η οποία έχει δημιουργηθεί στο Silicon Valley που βασίζεται στην επιστήμη. Είναι ένα νέο κίνημα, ξεπερνάει τον ανθρωπισμό και προσφέρει την αθανασία. Υπάρχει λοιπόν ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος στο να συνδυάσει κανείς την αμερικανική τεχνολογία με θρησκευτικές υποσχέσεις, η υπόσχεση της αθανασίας. Αυτή είναι μια νέα μορφή θεολογίας που έχει προκύψει και το δικό μου το ερώτημα προς τις ε, θρησκευτικές παραδόσεις είναι εσείς μπορείτε να προσφέρετε κάτι καλύτερο. Γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε όλοι σας ε, στην αίθουσα. Ήδη υπάρχει μία εκκλησία τεχνητής νοημοσύνης που την ίδρυσε αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε. Ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Apple παλαιότερα και αυτοί λένε ότι ο άνθρωπος ε, ακόμα δεν υπάρχει, αλλά θα έρθει κοντά μας με τη μορφή της ε, τεχνητής ε, νοημοσύνης. Θεός θα έρθει κοντά μας με τη μορφή της τεχνητής νοημοσύνης. Ε, υπάρχουν λοιπόν ανταγωνιστές και διερωτώ με τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτούς τους ανταγωνιστές. Well, thank you for, uh, for this presentation. Um, Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πρέπει να πω ότι ανοίξατε έτσι πολλά θέματα. Ε, έτσι ανοίξατε θέματα τα οποία χρήζουν συζήτησης. Θα διαβάσετε και τα κείμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι έχουμε μια μεγάλη ματιά, έτσι πιο ε, διαβριμένη. Μιλάμε για την πίστη, προσπαθούμε να μην επηρεαζόμαστε από, τον, από τις βιομηχανίες, πρέπει όμως να αντιληφθούν ε, πώς λειτουργούν αυτά τα δεδομένα, οι αλγόριθμοι, οι κώδικες ε, για να γνωρίζουν από εκεί και πέρα και πώς μπορούμε να έχουμε αυτή την ηθική ήδη στον αρχικό σχεδιασμό. Είναι δύσκολο λοιπόν, είναι περίπλοκο, ανοίξατε πάντως μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα τώρα να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Έχουμε τις πρώτες παρεμβάσεις από 5, λεπτών. Η Γιούλια Βίντοβιτς πρώτα εκπροσωπεί την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι καθηγήτρια βιοηθικής στο Παρίσι όπου διδάσκεται βοηθική οπότε ε, υπάρχουν πολλές προκλήσεις ό,τι αφορά την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης είναι και επίσημη εκπρόσωπο της ε, Σερβικής ε, Εκκλησίας έχετε το λόγο παρακαλώ ευχαριστώ θα μιλήσω γαλλικά σας ευχαριστώ όλους για αυτή την πρόσκληση είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντική. Θα μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για ένα θέμα τόσο σημαντικό σε πέντε λεπτά δύσκολο αυτό. Χρειάζεται έτσι να έχει κανείς ε, δυνατότητε σύνθεσης. Γι' αυτό λοιπόν θα επικεντρωθώ στους εξή άξονες. Πρώτα απ' όλα η σημασία των διαβουλεύσεων που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή και δεύτερον ε, δύο λόγια για το έγγραφο αυτό, το σχέδιο κειμένου σε ό,τι αφορά τι διαβουλεύσει. Όπω λέει και το έγγραφο τη διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, αυτέ οι διαβουλεύσει, οι δημόσιε, αυτέ οι συζητήσει, μόνο χρήσιμε μπορεί να είναι και να ενισχυθεί ε, το πνεύμα αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. Οι εκκλησίε ε, είναι το κατάλληλο έδαφο για τι συζητήσει αυτέ, μια και διαθέτουν μια μακρά και πλούσια παράδοση ε, συζητήσεων που σχετίζονται με τον άνθρωπο, το περιβάλλον του, το φυσικό του και πολιτιστικό του περιβάλλον και σε ό,τι μας αφορά σήμερα βεβαίως και τις σχέσεις ε, με την ηθική ε, και τη δημιουργία μεταξύ των οποίων και την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δηλαδή μια δημιουργία, έτσι, δεν είναι ο δημιουργός. Αυτές οι διαβουλεύσεις μπορούν να γίνουν ε, και να υπόκεινται υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι θετικό. Ε, το κείμενο όμως των ομάδα εμπειρογνωμών υψηλού επίπεδου και την τεχνητή νοημοσύνη ε, θεωρώ ότι πάει κάπως γρήγορα στο πώς ε, αντιμετωπίζει αυτά τα εξαιρετικά περίπλοκα ζητήματα. Θα αναφερθώ τώρα σε κάποιες σκέψεις που έχουν να κάνουν και με τη μέθοδο και την προσέγγιση αυτής της προβληματικής στο έγγραφο. Έχω την εντύπωση ότι το έγγραφο δεν λαμβάνει επαρκώ υπόψη το γεγονό ότι αντίθετα με την επιστημονική πρόοδο, η ηθική πρόοδο χρειάζεται χρόνο ο ρυθμός και η εφαρμογή σε μια ανθρώπινη κοινωνία είναι διαφορετική. Εάν θέλουμε να είναι πραγματική βιώσιμη και να μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή, η, η, ηθική εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών πρέπει να προέρχεται από, το, από τα κάτω, από την κοινωνία, η οποία είναι πολυπολιτισμική, είναι διαφορετική. Θα πρέπει από εκεί να οικοδομήσουμε με ανθρώπινο ρυθμό που δεν είναι αυτός των μηχανών Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, προσωμιώσουμε τον άνθρωπο με τη μηχανή και με τους ρυθμούς της. Πρέπει ο ρυθμός ζωής μας να είναι αυτοί που θα καθορίζουν τις ηθικές μας αξίες. Εμείς θα θέλαμε ουσιαστικά να παρακάμψουμε την, ε, τη σύνθετη διαδικασία λήψης ε, ηθικής θέσης. Η ηθική ακολουθούσε την τεχνολογική πρόοδο τώρα. Σήμερα όμως ε, για καλό σκοπό, για λόγους ασφάλειας στην πραγματικότητα, θα θέλαμε να βρεθεί μπροστά η ηθική από την τεχνολογία. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό όμως κάτι τέτοιο. Με βάση την δική μου παράδοση πρέπει να πω ότι μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση ή να υπάρξουν δηλαδή δύο, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητα βέβαια αλληλοαποκλεούμενες. Η ηθική από πάνω και η ηθική από κάτω. Όταν μιλάω για ηθική από τα πάνω είναι η προσέγγιση του εγγράφου. Έτσι. Δηλαδή καθορίζουμε κάποιες βασικές θεμελιώδεις ε, αξίες, ε, ηθικές ε, και δικαιώματα και συνέχεια τα εφαρμόζουμε. Το θέμα εδώ είναι ότι πρέπει να ξαναδούμε ε, τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των θεμελιωδών αξιών, των αρχών και των δικαιωμάτων. Πρέπει να μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Τι έχετε μπροστά Πρώτα, οι, οι τα θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις αρχές. Ποια είναι η θεμελιώδη αρχέ. και γιατί. Είναι σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση και πρέπει να αποτελεί μέρος του εγγράφου. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα σε ό,τι αφορά την ηθική από τα κάτω, αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση που νομίζουμε πως είναι και πλέον κατάλληλη. Δίνει σάρκα και πρεπει να αποτελει μερος του εγγραφου αυτο που αντιλαμβανομαι εγω τωρα σε οτι αφορα την ηθικη απο τα κατω αυτη ειναι μια διαφορετικη προσεγγιση που νομιζουμε πω ειναι και πλεον καταλληλη δινει σαρκα και οστα στο όλο εγχείρημα. Θα βασιστούμε στην εμπειρία, στις πολλαπλές εμπειρίες, ποικίλε εμπειρίες που προέρχονται από διάφορους τομείς που πλήττονται ή που επηρεάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη και την εφαρμογή της. Αυτό θα μας επιτρέψει ε, να, να έρθουμε στον πραγματικό διάλογο, να δημιουργήσουμε μια συζήτηση που θα αφορά όλο και περισσότερους πολίτες, συζητήσεις που θα έχουν πραγματικό νόημα, διότι στην πρώτη μου ανάγνωση του εγγράφου αναρωτιόμουν σε ποιον απευθύνεται τελικά το έγγραφο αυτό. Ο κανόνα λέει ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε σε όλου, ουσιαστικά είναι σαν να μην μιλάμε σε κανέναν. Να δώσω ένα παράδειγμα. Διαβάζοντα τον έγγραφο, έβλεπα μόνο κάποιε γενικότητε στο τι εννοούμε όταν λέμε ανθρώπινο όν, χωρί να λαμβάνεται υπόψη η περιπλοκότητα τη ανθρώπινη διάσταση. Τη βιολογική του, φυσιολογική, ψυχολογική, κοινωνική, πνευματική διάσταση. Και για την ελευθερία του βέβαια. Η ελευθερία του ανθρώπου καθορίζεται με βάση την επιλογή πώς συνδέεται η αυτονομία με την ελευθερία, την του ανθρώπου, παραδείγματο χάρη. Πολύ σημαντικά θέματα ε, που είναι στο κέντρο της χριστιανικής ανθρωπολογίας και μπορεί να πάει σημαντική συνεισφορά εδώ. Αυτό που εγώ θεωρώ ότι λείπει στο έγγραφο αυτό είναι η διασύνδεση μεταξύ της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, της θεολογικής και της πολιτικής της ηθικής πολιτικής και της πρακτικής σοφίας. Θα πρέπει λοιπόν οι υπάρχουσες ηθικές ε, να είναι ε, πιο ισορροπημένε. Υπάρχει η, ηθική του Αριστοτέλη και του Κάντα από την άλλη, υπάρχει από τη μία η πιο έτσι ε, ωφελημιστική ε, ηθική, ε, άλλο η τεχνική, άλλο η νομική, ε, υπάρχει η υποκρατική ηθική την οποία ακολουθούν και οι μουσουλμανικοί και οι καθολικοί πρέπει να έχουμε κατά νου τις αξίες που συνδέονται με το πρόσωπο όμως, τον άνθρωπο απευθείας Μίλησαμε για αξιοπρέπεια, ανθρώπινη αξιοπρέπεια προηγουμένω και μια ηθική που να επικεντρώνεται στην ε, επιφυλακτικότητα. Ε, δεν μου αρέσουν οι γενικολογίε, αλλά συνήθω δίνεται έμφαση στι στις προσωπικέ, στι ατομικέ αξίε, στην αγγλοσαξονική προσέγγιση, χωρί να θέλω να γενικεύσω. Είναι λίγο καρικατούρα βέβαια αυτό, αλλά θέλει προσοχή Και βεβαίως υπάρχουν οι βασικές τέσσερις αρχές της, του σεβασμού της αυτονομίας, του, του να κάνει κάποιος το καλό, του να μην κάνει το κακό, της αυτονομίας. Όλα αυτά δεν σχετίζονται απαραίτητα μεταξύ τους και ιδιαίτερα όταν οι αρχές αυτές οι ηθικές αντιφάσκουν σε ό,τι αφορά την τεχνική λύση. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, μιας και βασιζόμαστε σε αυτές τις αρχές. Για το σημείο αυτού λοιπόν θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς η ομάδα διαβούλευσης εξετάζει ε, παίρνει θέση σε ό,τι αφορά το γεγονό ότι υπάρχουν δράστε, παράγοντε με διαφορετικά συμφέροντα που αντιλαμβάνουν διαφορετικά αυτέ τι αρχέ. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, θα ήθελα επίση να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο που λέει ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε τη, το, το, τη σχέση μεταξύ των διαφόρων ηθικών. Θα πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τι διάφορε ηθικέ. Την ηθική τη έρευνα, την πολιτική ηθική, την οικονομική ηθική, την φιλοσοφική και θεολογική ηθική. Το πώ η κάθε μία από αυτέ αντιλαμβάνεται, εξηγεί ε, την τεχνολογική και επιστημονική ε, πρόοδο για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το, το καλούπι της ε, κατανάλωσης και του ανταγωνισμού. Αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα με μια κριτική προσέγγιση πολυσχηδής που θα βασίζεται σε, στην ακαδημαϊκή παιδεία όπου θα, θα συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι κλάδοι η επιστημονική. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τίξατε πολύ σημαντικά θέματα ε, και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που έχουν προκύψει και που πρέπει να εξετάσουμε. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο. Θα έχουμε μετά στο τέλος ε, χρόνο για ερωταπαντήσεις. Ντομινίκ Λαμπέρ, πρόσωπος των Καθολικών, εκπροσωπεί την Καθολική Διάσκεψη ε, Επισκόπων, με Επισκόπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσης φιλόσοφος ε, και ε, φυσικός, τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ναμούρ, Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ που έρχονται στη συζήτηση αυτή. Θα δώσω έμφαση σε τέσσερα σημεία, σε τέσσερις κατευθύνσεις γραμμέ που προέρχονται από την καθολική παράδοση που θα μπορούσαν να βοηθήσουν για να γίνει μια αξιολόγηση των αναπτύξεων, τη ανάπτυξη τη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη, ε, στι ευρωπαϊκέ μα κοινωνίε. Το πρώτο σημείο είναι η κρίσιμη αναφορά στο πραγματικό ανθρώπινο «ον» που δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι είναι μια συσκευή, ένα πράγμα, κάτι τεχνητό. Το δεύτερο είναι η αναγκαιότητα να διαφυλάξουμε το ανθρώπινο περιεχόμενο ε, και τους σκοπούς των διαφορών πράξεων. Ε, η, επίσης, τρίτον, η απέτηση του να διαφυλάξουμε την ε, αδερφοσύνη την παγκόσμια στην ανθρωπότητα και να διαφυλάξουμε επίσης το κοινό μας σπίτι, το κοινό μας οίκο και το κοινό καλό. Σε ό,τι αφορά τώρα το ανθρώπινο το πρώτο στο οποίο αναφέρθηκα, που δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι ε, ένα αντικείμενο. το ανθρώπινο «ον» είναι ένα σημείο αναφορά, το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει κανεί. Θέλουμε να πούμε ευθύ εξ αρχή ότι η ηθική αξιολόγηση τη τεχνητή νοημοσύνη και άλλων αυτόνομων συστημάτων πρέπει να βασίζεται στη μια σαφή εικόνα του τι είναι ο άνθρωπος και ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ανθρώπινου όντως και των μηχανών. Πολύ συχνά η, το λεξιλόγιο, η ορολογία έρχεται να αλλοιώσει την ε, αξιολόγηση αυτή. Υπάρχει μια ταύτιση και μια σύγχυση σε ό,τι αφορά το αντικείμενο και τον άνθρωπο. Η προσωμείωση, η, η αναπαράσταση ανθρωπίνων συμπεριφορών ε, δημιουργεί αυτή τη σύγχυση. Και αυτό οδηγεί σε πολλές, πολύ μεγάλες και νομικέ, αλλά και ηθικές ανησυχίες. Ένα μηχάνημα δεν μπορεί πραγματικά να αποτελέσει νομικό ή ηθικό πρόσωπο. Δεν, η συμπεριφορά του δεν βασίζεται ε, σε πραγματική σκέψη και δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο ένα αντικείμενο για κάποιες πράξεις και ούτε ένας άνθρωπος μπορεί να βασίζεται να, τον, να τον μόνο με βάση την απόδοσή του η οποία να ποσοτικοποιείται. Πρέπει, όταν σεβόμαστε τον, τον άνθρωπο πρέπει να σεβόμαστε και το ρυθμό του. Είναι σημαντικό λοιπόν κατά την ηθική αξιολόγηση της τεχνητής νοημοσύνης να μην θεωρήσουμε ότι η ανθρωπότητα πρέπει να ακολουθεί τους ρυθμούς των ρομπότ. Ορισμένες φορές είναι σημαντικό και είναι και πιο ασφαλές να σεβαστούμε αυτό το ρυθμό του ανθρώπου και να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί η μηχανή να επιβάλλει την ταχύτητά της, το ρυθμό της στην ανθρώπινη κοινωνία. Θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ το θέμα αυτό του χρόνου. Είναι από μια από τις βασικές σκέψεις του κεκτημένου του καθολ... της Καθολικής Εκκλησίας και υπάρχουν πολλές έρευνες στο παρελθόν επ' αυτού, του Henry Gilliam παραδείγματος χάρη, ε, ανάγκη επίσης το να διαφυλάξουμε το, το ανθρώπινο περιεχόμενο και τον σκοπό των δράσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία, μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να παραμείνει στην υπηρεσία του συνόλου τη ανθρωπότητα, χωρίς να ξεχνάμε τι ανθρώπινε και κοινωνικέ ε, και κοινωνικούς στόχους θέλει προσοχή ήδη από, την, από των αλγορίθμων έως τη χρήση τους. Όταν λοιπόν μοιράζομαστε την εξουσία με τις μηχανές, όταν υπάρχει εξουσιοδότηση, θα πρέπει να είναι σαφής ποιος, ποιο είναι, ποιος είναι ο σκοπός των ανθρώπων. Όταν μιλάμε για προστασία των ανθρώπων, πρέπει να έχουμε αξιόπιστα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και να υπάρχουν νομικές απαιτήσει να μπορούμε να εξηγήσουμε τις διαδικασίες αυτές που ελέγχει ο αλγόριθμος όταν μιλάμε για λήψη αποφάσεων αυτοματοποιημένη. Το να υπάρχει έλεγχος από τον άνθρωπο της τεχνής νοημοσύνης είναι κρίσιμο και για τα συστήματα τα οπλικά. Η Καθολική Εκκλησία θέλει να προτείνει απαγόρευση των οπλικών συστημάτων όταν ο άνθρωπος είναι εκτός της χρήσης αυτής. Διότι υπάρχει κίνδυνος παραβίασης ε, των διεθνών αρχών του, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Να μην έχουμε τη δυνατότητα πλέον πολιτικής δράσης και να οδηγήσει βεβαίως αυτό και στο θάνατο ανθρώπων. Επίσης υπάρχει η, το σημαντικό αίτημα της, εν, ανθρωπότητας και της αδελφοσύνης. Πρέπει να έχουμε αυτήν την παγκόσμια αδελφοσύνη και εδώ αναφέρομαι σε αυτά που είπε και ο Πάπας Φραγκίσκος ε, ορισμένες φορές αυτή η αδελφοσύνη πλήττεται από, από τις ε, διακρίσεις ε, που προκύπτουν στους αλγόριθμους και λόγω τεχνικών κενών, γυρογμών που έχουν να κάνουν με διαφορετικές δυνατότητε πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους. Αυτή λοιπόν η αδελφοσύνη ε, προϋποθέτει ότι θα πρέπει να υπάρχουν εργα, ε, εργαλεία τεχνητή νοημοσύνη που αναλαμβάνουν υπόψη και τα ατόματα με ειδικέ ανάγκε. Ε, αυτή η ηθική ζητάει, μα ζητάει να σκεφτούμε την αναγκαιότητα να έχουμε συστήματα μακροπρόθεσμα και να υπάρχουν και άνθρωποι με σάρκα και οστά στα συστήματα αυτά. Πρέπει να μπορεί να υπάρχει μια διάδραση πραγματική, πρόσωπο με πρόσωπο η ρομποτοποίηση δεν πρέπει να ε, γίνεται λειπτή ως ότι το πραγματικό σώμα το βιολογικό δεν έχει πια σημασία για να περιθάλψει παραδείγματος χάρη τους ηλικιωμένους ε, δεν μπορεί αυτό να το κάνει μόνο ένα μηχάνημα ή μια οθόνη μας δείχνει ε, το σκοτεινό πρόσωπο του διαδικτύου ότι ορισμένε φορές η τεχνολογία μπορεί να χωρίσει τους ανθρώπους και τα έθνη θα πρέπει λοιπόν να γίνει σεβαστή και η ιδιωτικότητα των ανθρώπων και πρώτα απ' όλα οι πιο ευάλωτοι εξ αυτών θα προστατευθούν από τις ε, κυβερνοεπιθέσεις, ε, την ε, παρενόχληση στο διαδίκτυο. Αν θέλουμε να, επανεκοδομήσουμε τα αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα λύθης, να μπορούμε να γράψουμε κάποιες πληροφορίες στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με τα συστήματα data mining. Να διτρήσουμε, το να διτρούμε κάποια στοιχεία που αφορούν ανθρώπους σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε την εξέλιξη του ανθρώπου και το, ο άνθρωπος αυτός ουσιαστικά εγκλωβίζεται για πάντως ψηφιακό του προφίλ. Αυτή η αλγοριθμική ε, αιωνιότητα παγώνει τον άνθρωπο σε ένα συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δεν δέχεται ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται και ότι το ανθρώπινο μπορεί ε, να συγχωρεθεί για κάτι. Και τέλος, η διαφορά ε, η προστασία της, του κοινού μας οίκου και του κοινού καλού. Γίνεται ιδιαίτερα, ιδιαίτερη αναφορά στο κοινό καλό, στο, στα κοινά αγαθά. Οι νέες τεχνολογίες, τα, τα ρομπότ πρέπει να είναι στο συμφέρον του κοινού καλού της κοινωνίας και να μην αναπτύσσεται μόνο προς όφελος μικρών ομάδων. Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης στα πλαίσια της προοπτικής αυτής πρέπει να σέβεται και το περιβάλλον τα πρόσωπα, και οι χώρες που παράγουν αυτά τα χημικά προϊόντα ε, για να παρασκευάσουν αυτές οι συσκευές ξέρουμε ότι προέρχονται συχνά από αλυσίδες ε, που ε, εκμεταλλεύονται παιδιά ή πολύ φτωχούς εργαζόμενους. Υπάρχουν και περιβαλλοντικές, περιβαλλοντικά ζητήματα που να ληφθούν υπόψη. Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά ποιοι είναι αυτοί που θα χάσουν την εργασία τους λόγω της νέας αυτής της τεχνολογίας και πώς θα τους προσφέρουμε νέες δυνατότητες ε, να μπορέσουν ε, να συνεχίσουν να εργάζονται. Τελειώνοντας να πω ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προτείνουμε μια ηθική αξιολόγηση της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών των σχετικών με βάση αυτές τις κατευθύνσεις γραμμές σεβασμός όλων των διαστάσεων του ανθρώπου και του κοινού καλού, του κοινού οίκου και των πολιτών αυτού. Πρέπει να υπάρχει μια, μια αρχή ανθρωπολογικής συνοχής. Να αναπτύξουμε τις, τις τεχνολογίες της τεχνητής νοημοσύνης σεβόμενοι και ενισχύοντας όλους τους ανθρώπους λαμβάνοντας υπόψη την βιολογική του, την κοινωνική του διάσταση, το πνευματικό του βάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και φαντάζομαι όλοι θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να σεβαστούμε τις ανθρώπινες αξίες και να ορίσουμε ε, παγκόσμιες ε, αξίες ε, που να τις σεβόμαστε όλοι. Ίσως να μην έχουμε όλοι τις ίδιες, αλλά πιστεύω ότι οι ανθρώπινες αξίες είναι κοινέ, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι από αυτού. Και τώρα θα ακούσουμε την κυρία Σουάντο Ονισέλκα, εκπρόσωπο των μουσουλμάνων, δάσκαλα στη Φινλανδία. Είναι επίσης ε, ειδική ε, στην ομάδα στο Ελσίνκι. Έχει εργαστεί για την Ισλαμική εκπαίδευση ε, στην Φινλανδία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που οργανώνετε αυτό το σεμινάριο γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μοναθέστε κάτι πολύ δύσκολο, το να μιλήσω εκ μέρους των μουσουλμάνων γιατί ξέρουμε ότι μιλάμε για 1,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αν δούμε την Ευρώπη είναι 40 εκατομμύρια και αν δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 19 εκατομμύρια. Όταν μιλάμε για τις ηθικές επιφυλάξεις, αυτό δεν είναι τίποτα το καινούργιο στη μουσουλμανική κοινότητα, γιατί αντιμετωπίζουμε πολύ, ε, πολλές διακρίσεις, ξενοφοβία, ισλαμοφοβία, αυτά τα τελευταία χρόνια. Και τα σημαντικότερα θέματα είναι αυτά και τα οποία έχουν τεθεί. Όσον αφορά λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη, για μας τεχνητή νοημοσύνη είναι ε, ανθρωπογενής. Αν δούμε δηλαδή πόσοι άνθρωποι έχουν προκαταλήψεις έναντι των μειονοτήτων και οι αλγόριθμοι ε, δεν στερούνται προκαταλήψεις. Θα αναφέρω κάποια παραδείγματα. Ε, σχετικά πρόσφατα, παραδείγματος χάρη Υπάρχουν διάφορες ε, εφαρμογές για την υγεία ε, που συγκεντρώνουν δεδομένα για έναν άνθρωπο. Είναι εφαρμογές ε, για άντρες και για γυναίκες, αλλά δεν δεν έχουν συγκεντρώσει στοιχεία για την, τον, την έμεινη ρίση των γυναικών που είναι σημαντική για τις γυναίκες αλλά όχι φυσικά για τους άντρες. Και αυτό είναι ένας παραδείγματος χάρη αλγόριθμος. Ε, αν δούμε και τις κάμερες που υπάρχουν σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, το μοβ δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλα χρώματα. Δεν είναι τόσο συγκεκριμένο όπως άλλα χρώματα και ποιος υποφέρει τελικά από αυτό είναι οι άνθρωποι που έχουν ε, πιο σκούρο δέρμα. Ή όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να ρίξουμε ένα βλέμμα γύρω μας και να σκεφτούμε τι είδους προκαταλήψεις έχουμε ο ένας για τον άλλον. οι κάμερες ε, δεν μπορούν να τα καταφέρουν τόσο καλά ε, με την ανάλυση των χρωμάτων, ε, αλλά στις φωτογραφικές κάμερες τα μάτια μοιάζουν να είναι ροζ, φούξια. Στη Φινλανδία, εγώ είμαι εκπαιδευτικός και θα μιλήσω βέβαια για το σχολείο, Αναφέρθηκε ήδη ότι το σχολείο είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπιστούν κάποια ηθικά προβλήματα που συζητάμε. Στο ε, σχολικό πρόγραμμα της Φινλανδίας υπάρχει κριτική σκέψη που εντάσσονται μέσα στα σχολικά προγράμματα. Νομίζω σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει και τα δύο να τα περιλαμβάνουμε όλες οι χώρες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να μπορούν να προστατεύονται και γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τις ε, θεωρίες των αλγορίθμων και όταν είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μην ξέρουν καν τη λέξη αλγόριθμος. Και κάτι άλλο. Τώρα τα σχολεία είναι χώροι marketing για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δούμε λιγάκι τις αναλύσεις δεδομένων, τα σχολεία ε, εξοπλίζονται όλο και περισσότερο με μηχανές ε, που συγκεντρώνουν δεδομένα και τι γίνεται μετά με αυτά τα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα ισχύουν και κάτω από το πρίσμα των μειονοτήτων. Μήπως μετράνε στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για την πλειοψηφία ή μήπως συγκεντρώνουν πληροφορίες που να είναι σημαντικές και για τις μειονότητες. Όσον αφορά τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης, την Παρασκευή ε, είδαμε το τι μπορεί να συμβεί στα χέρια των παιδιών. Ξέρουμε τι συνέβη την Παρασκευή στη Νέα Ζηλανδία αυτή η ε, απεχθής ε, επίθεση. Εγώ διδάσκω μόνο λίγες ώρες την εβδομάδα. Διδάσκω μαθηματικά στην 7η τάξη και ξέρω βέβαια ότι οι μαθητές μου διαβάζουν τις ειδήσει, ε, μπαίνουν στο διαδίκτυο και αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα για το πώς η τεχνητή νομοσύνη επηρεάζει κάθε μέρα τη ζωή των παιδιών μας. Έκανα πολλές ερωτήσεις στους μαθητές, τους ρώτησα τι είδους ειδήσει ε, διαβάζετε αυτά ε, μάλλον πρέπει να υποστηρίξω ότι και στη μουσουλμανική κοινότητα βλέπουμε ότι οι ειδήσει δεν είναι πάντα ιδιαίτερα θετικές, ε, δεν διαφέρουν πολύ από τον δυτικό κόσμο. Η παροχή ειδήσεων, μήπως ε, αυτή οδηγεί στο να γινόμαστε λιγότερο άνθρωποι. Ε, πώς μας επηρεάζουν όλα αυτά, πώς σκεφτόμαστε για τους συνανθρώπους μας. Γι' αυτό το λόγο η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και κατανόησης της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ σημαντική, γιατί διαμορφώνει τις απόψεις μας και θα πρέπει ε, να εντάσσεται στις ικανότητες όλων ως πολιτών. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο οι νέοι. Υπάρχουν και πολλοί ενηλίκες οι οποίοι θα επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, θα επηρεαστεί ο κόσμος μας με διάφορους τρόπους. Ε, κάποια επαγγέλματα ε, θα εξαφανιστούν, θα εμφανιστούν άλλα. Και πώς θα αντιμετωπίσουμε εκείνους τους ενήλικες που χρειάζονται νέα εκπαίδευση για να μπορέσουν να ζήσουν σε αυτή την Ήπειρο. Σε πολλά μέρη του κόσμου η τεχνητή νομοσύνη αντιμετωπίζεται ως κάτι πολύ επικίνδυνο γιατί πολλοί θεωρούν ότι τους αφαιρεί ε, τα επαγγέλματά τους. Τελικά η τεχνητή νομοσύνη ε, μας κάνει πιο ανθρώπους. Ελπίζω να συμβαίνει αυτό. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι χωρίς ηθικές κατευθυντήριες γραμμές ε, τα δεδομένα δεν μας καθιστούν πιο σοφούς. Πραγματικά χρειαζόμαστε ηθικές κατευθυντήριες γραμμές. Είχα κατά νου το σοφισμό. Αν δείτε λιγάκι το θέμα έτσι κάτω από το πνεύμα των φιλοσόφων, έχουμε τρία διαφορετικά τετρα... τρεις κύκλους. Ε, απ' έξω είναι ο Ισλαμικός νόμος, όπως και τα ε, τεχνητά δεδομένα. Μετά πάμε στην εσωτερική πίστη είναι η ανάλυση των δεδομένων και στο τέλος υπάρχει η μαρίφα όπως λέμε ε, κάτι το ιερό που θα μπορούσε να είναι η ηθική και ο τρόπος ε, με τον οποίο λειτουργεί η Τάρικα είναι ο αλγόριθμος που μας φτάνει ως το τέλος. Ελπίζω ε, ως άνθρωποι να έχουμε ελεύθερη βούληση όταν θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη θεωρία των αλγορίθμων και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα ε, για να συζητήσουμε. Θα θέλω να δώσω τον λόγο στην κυρία Ντεκάιζερ, η οποία είναι εκπρόσωπος ε, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ουμανιστών. Υπήρξε ευρωβουλευτής για πάρα πολλά χρόνια. Ε, θεωρώ ότι η άποψή της είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, την φίλη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναρωτηθεί κανείς ποιος θα είναι ο κοινωνικός έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης. Μία από, ένας από αυτούς είναι ε, ποια είναι τα καθήκοντα τα οποία τώρα ε, εκτελούν άνθρωποι μπορούμε να δεχθούμε να τα αναλάβουν μηχανές. Αυτό το ερώτημα τέθηκε σήμερα. Βλέπουμε πολύ, ότι πολύ γρήγορα αυτό μας οδηγεί σε φιλοσοφικά, ηθικά ζητήματα, ζητήματα ηθικής. Έχουν συζητηθεί αυτά σε πολλές κριτές γραμμές για την ηθική. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτές τις γενικές συστάσεις. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανθρωπιστών εμπνεύστηκε από αυτές στο μανιφέστο της για τις εκλογές του 2019. Ε, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο τύπος της κοινωνίας με τεχνητή νοημοσύνη ε, στην οποία μπαίνουμε δημιουργεί νέους κινδύνους κίνδυνοι οι οποίοι ορισμένε φορές, ορισμένες φορές έχουν να κάνουν με την ίδια δομή, την ίδια τη δομή αυτών των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Το έχουμε αξιολογήσει αυτό, το έχουμε ταξινομήσει, τα έχουμε ε, αποκλείσει. Γι' αυτό θέλω να μιλήσω σήμερα, διότι το όριο στο τι μπορούμε να δεχτούμε δεν έχει να κάνει και δεν πρέπει να έχει να κάνει μόνο με το πολιτικό με το ηθικό ζήτημα, με το θέμα της ισότητας, ή το νομικό επίπεδο μάλλον, έχει να κάνει και με το ποιο είναι το επίπεδο κινδύνου, το ποσοστό κινδύνου που μπορεί να αποδεχτεί μια κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο αυτό, διότι εξέτασα το σχέδιο του κειμένου, δεν έχω λάβει την τελευταία εκδοχή βεβαίως από το πάνελ εμπειρογνωμών κυρία Μέτσιγκερ, ε, για τα ζητήματα ηθικής, βρήκα ότι το κείμενο αυτό, το είπατε κι εσείς δηλαδή, ε, ότι το κείμενο αυτό είναι κάπως τρευλό, ε, δηλαδή πάει πολύ προς το τεχνολογικό σκέλος, οδηγεί σε μια επιχειρηματολογία οικονομικού τύπου, ε, από ό,τι βλέπω στο πάνελ αυτό υπήρχαν πολλοί οικονομικοί παράγοντες, οπότε φυσιολογικό είναι να ε, πάει προς τα εκεί το κείμενο. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση, κυρίως, είναι ότι δεν υπήρχε καμία πραγματική αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε και καμία επιλογή δεν δίνεται στην κοινωνία. Εάν το θέλουμε αυτό ή αν δεν το θέλουμε, παραδείγματος χάρη. Όχι βάσει κάποιας ηθικής αξίας, όχι βάσει κάποιας νομικής προσέγγισης, αλλά με βάση αυτό που εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να, να δεχτούμε ως αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Εγώ βεβαίω υπερασπίζομαι την τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω ότι θα κάνουμε πραγματικά καταπληκτικά πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά θέλω να γνωρίζω ορθολογικά τι συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή, και το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος. Δημιουργούμε κάθε μέρα μια κοινωνία όπου ο κίνδυνος είναι αναπόφευκτος. Η αξιολόγηση κινδύνου γενικότερα, η πρόληψη και η διαχείριση έχουν αποτελέσει αντικείμενο σε διάφορα προγράμματα πλαίσιο έρευνας της Ένωσης, ε, ενός οπλοστασίου ε, μέσων ε, σε ό,τι φορά την, ε, το πυρηνικό τομέα, στην πληροφορική, αλλά και στην νομοσύνη. Και εγώ προσωπικά το έχω δοκιμάσει. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ ήμουν ειδική στο πρόγραμμα Drive τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεκαετία του 90 και συμμετείχα σε εμπειρίε ό,τι αφορά οχήματα που θέλαμε να είναι αυτόνομα. Υπήρχε ένας, ένα αυτόματο σύστημα οδήγηση ήδη από τότε στι 100 χώρε. Και η σύγκρουση μεταξύ της λογικής του ανθρώπου και της λογικής του αυτόματου οδηγού ε, είναι μια σύγκρουση την οποία τη ξαναβρήκαμε μετά και στα αεροπλάνα ε, όπου υπάρχουν ε, πιλότοι με τεχνητή νοημοσύνη στην δεκαετία του 90 είχαμε τα Airbus 300, τα Airbus 320 είχαμε την καταστροφή στο Σαντοντήλ και, οδηγη, και οδηγηθήκαμε στην καταστροφή αυτή λόγω τη σύγκρουση μεταξύ τεχνητή νοημοσύνη και τη λογική τη ανθρώπινη. Και νομίζω πω κάτι τέτοιο τελικά συνέβη και με την Ethiopian Airlines πρόσφατα, με τα Boeing αυτά τη νέα γενιά. Και αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτέ είναι επιλογέ μια κοινωνία. Έχουμε μια παράδοση. Έτσι, μπορεί να είμαστε λίγο πίσω στον ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είμαστε πίσω σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της τεχνολογίας, την αξιολόγηση του κινδύνου, όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι όταν σχεδιάζουμε νέες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και λέγεται αυτό στις γραμμές, πρέπει να είναι συμμετοχική η διαδικασία με διάφορους παράγοντες από το σχεδιασμό έως την εφαρμογή. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε ακόμα περισσότερο είναι ότι ακόμα και αν το προσέξουμε, προσέξουμε πάρα πολύ πώς σχεδιάζουμε αυτό το τεχνολογικό εργαλείο, πάντα θα υπάρξουν προβλήματα, δυσλειτουργίε, ατυχήματα. Θα υπάρξει δυνατότητα να δούμε τι γίνεται στην πράξη, να, να, να αξιολογήσουμε τις εμπειρίες, να συλλέξουμε δεδομένα. Για την ώρα δεν συλλέγονται αυτά τα δεδομένα. Γίνεται μια συλλογή, παραδείγματο χάρη στο μέρο τη αεροναυπηγική, και εκεί έχουμε ατυχήματα που αφορούν τεχνητή νοημοσύνη. Στον πυρηνικό τομέα επίσης, στα πυρηνικά εργοστάσια. Και εκεί συμβαίνουν ατυχήματα τα οποία καταγράφονται, τα αναλύουμε και ε, τα επεξεργαζόμαστε. Αυτό που δεν έχουμε όμως είναι μια ορατότητα του τι έχουμε στη διάθεσή μα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανθρωπιστών ζήτησε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Διότι με την εξέλιξη αυτών των νέων εργαλείων, ε, είπαμε ότι πρέπει να μπορούμε να εξηγήσουμε του αλγόριθμου. Εντάξει. Αλλά ποιο δεν ξέρει σήμερα ότι σε αυτά τα εργαλεία νέας, ε, νέας γενιάς είναι όλο και πιο ασαφές το ζήτημα. Δεν είναι μόνο οι αλγόριθμοι. Είναι πώς να πάνε η χώρα επεξεργασία ε, των δεδομένων στα διάφορα δίκτυα που μας συνδέουν να καταλάβουμε ακριβώς ότι τα λάθη έχουν να κάνουν με το γεγονό ότι οι απαντήσει ε, διέπονται από τον νόμο των πιθανότητων. Και πάντα υπάρχει ένα ποσοστό λάθου. Όλα αυτά θα πρέπει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπειρία, με την εμπειρία που έχει, έχει δημιουργήσει υπηρεσίε για τόσα πράγματα. Ε, είναι ένα διακύβευμα σημαντικό. Υπάρχει το θέμα τη ηθικής, αλλά όταν θα έχουμε κάτι τέτοιο, αυτό το εργαλείο, θα μπορούμε να πούμε τότε στην κοινωνία, ξέρετε, το επίπεδο κινδύνου διότι η επιλογή μιας κοινωνίας γίνεται και με βάση το ποιο είναι το ποσοστό κινδύνου που μπορούμε να δεχτούμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και στοιχεία ψυχολογικά, πολιτιστικά. Δέκα νεκροί στον τομέα της δημιουργίας και δέκα νεκροί στον, στον, τομέα της πυρηνικής ενέργειας δεν είναι το ίδιο. Όταν υπάρχουν δέκα νεκροί λόγω πυρηνική ενέργεια, κλείνει ο πυρηνικό εργοστάσιο. Εργοστάσιο είναι διαφορετική η ευαισθησία, εντάξει. 10 νεκροί όμως ε, με οχήματα που είναι ε, που προκύπτουν από αυτόματη οδήγηση, αυτό είναι παραδεκτό. Μιλάμε για 10 νεκρούς όμως από απλό ατύχημα, δυστύχημα αυτοκινηστικό, τότε δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Λοιπόν, εγώ ζητώ να φτάσουμε σε μια κοινωνία που θα μπορεί να αξιολογεί το κίνδυνο και έτσι να μπορέσει να ελέγξει, να δαμάσει την τεχνητή νοημοσύνη ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία. Διότι έτσι μπορεί κανείς να πάρει τις αποφάσεις του αμερόληπτα, απαντώντας και σε πράγματα που ελέγχθησαν νωρίτερα πολύ σωστά. Well, you help me give the floor now, uh, since... Έχει εξειδικευτεί ε, ή είχε εξειδικευτεί σε θέματα ε, διαιτησιών ε, πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Ο συνάδελφός μου κύριος Φόξ και νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, πολύ καλύτερη από αυτή που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και θα ήθελα να ε, του δώσω την ατότητα να επισημάνει ορισμένα θέματα και αυτά που ελέγξα να τα συσχετίσει και με την ε, εκθεσή μας. Άσλη, συγχαρητήρια και έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Εύα, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε που φιλοξενείτε σήμερα τη συζήτηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μέχρι τώρα και ευχαριστώ πολύ για όλα όσα ελέγχθησαν. Ως Βρετανός είναι βέβαια πάρα πολύ ενδιαφέρον το να έρχεται κανείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μιλάει για κάτι άλλο και όχι πια για τον Brexit. Γιατί ασχολούμεθα με τα κοινά, μερικοί εξημών Πιστεύω για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής ε, των ε, ανθρώπων μας κατά τον 10 ο αιώνα, αυτά είπε ο Μπεντζαμιν τιζραηλη Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι ενθουσιασμένος ε, ε, με την τεχνητή νοημοσύνη και είμαι αισιόδοξο για το μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλέ τεχνολογίε οι οποίοι ε, διαχρονικά έχουν αλλάξει την ανθρώπινη ζωή, την έχουν κάνει καλύτερη και ε, εκεί που βρισκόμαστε τώρα είναι το σημείο όπου βρισκόταν η ανθρωπότητα πριν από 300 περίπου χρόνια, την εποχή του ατμού. Τότε είχαμε αυτές τις πρωτόγονες μηχανές ε, τότε ο ατμός χρησιμοποιείται μόνο στα ορυχεία. Ξεπέρασαν από τότε 300, 300 ε, χρόνια και είχαμε μετά ε, τις ατμομηχανές που διέσχιζαν τις υπήρους. Θεωρώ λοιπόν ότι η τεχνητή νομοσύνη είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ αρχικό στάδιο και μπορούμε να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τα επόμενα 200 χρόνια πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα με αυτά που είπε η κυρία Ντεκάιζερ σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων. Πρέπει να αξιολογούμε τους κινδύνους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μετά από 20 χρόνια τα περισσότερα οχήματα θα είναι αυτόνομα. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι κάθε φορά που θα υπάρχει ένα ατύχημα και θα σκοτώνεται κάποιος από ένα αυτόνομο όχημα, ε, θα ε, εξαγριώνονται όλοι πολύ περισσότερο από αυτό που πραγματικά του αξίζει αναλογικά. Γιατί, Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι τέλεια και θα σκοτώνονται κάποιοι άνθρωποι, αλλά κατά την άποψή μου θα χάνουν τη ζωή τους πολύ λιγότερη από το να επιτρέπουμε στους ανθρώπους ε, να συνεχίσουν να οδηγούν τα αυτοκίνητα. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε το θέμα και πρέπει να αξιολογήσουμε ε, ορθολογικά τους κινδύνους. Και μερικές φορές αυτό δεν το καταφέρνουμε καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρτε τους, ε, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Υπάρχει μια πολύ αυστηρή διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τους επιστήμονες που αναλύουν αν προϊόντα είναι καλά και αφού εγκριθούν μετά το κοινοβούλιο λέει όχι δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσουν αυτά, ε, δεν μας αρέσουν έτσι απλά και όχι γιατί υπάρχουν κάποια επιχειρήματα. Και αυτό το βιώνουμε ακούμε συνεχώς. Η πολιτική πολύ συχνά δεν είναι πολύ καλή στο να επιχειρηματολογούν με βάση τη λογική. Στη δική μου την έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη ε, τοποθετηθήκαμε θετικά. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένα περιβάλλον όπου γίνονται επενδύσει, όπου η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας, ε, την υγεία μας, ε, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης που δεν υπάρχουν και που θέλουμε να ελπίζουμε θα μας δώσουν και περισσότερο χρόνο για αναψυχή, πολύ περισσότερο από ό,τι κατά το παρελθόν. Πολλοί βουλευτές θα πούν ναι, αλλά θα καταστραφούν ε, θέσεις απασχόλησης. Βεβαίως και θα συμβεί αυτό, όπως και η ατμομηχανή κατέστρεψε πολλές θέσεις απασχόλησης, όπως και μηχανές εσωτερικής καύσης, όπως συνέβη και με τους υπολογιστές. Σας λέω λοιπόν ότι ανταυτού όμως θα δημιουργηθούν πολύ περισσότερες θέσεις από αυτές που θα χαθούν και είναι σημαντικό να αγκαλιάσουμε αυτή την τεχνολογία με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όταν θα λειτουργούν αυτοί οι αλγόριθμοι. Όπως είπε και ο καθηγητής κ. Λαμπέρ, θα πρέπει να παραμείνουν στην υπηρεσία των ανθρώπων και να ελέγχονται, συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την άποψη. Όμως δεν πρέπει να προχωρήσουμε πολύ αργά. Κάποιος είπε ότι προχωράμε πολύ γρήγορα. Ε, καθηγητής Βίντοβιτς νομίζω είπε ότι προχωράμε πολύ, αργά, πολύ γρήγορα. Με συγχωρείτε. Όχι, δεν προχωράμε τόσο γρήγορα γιατί παραδείγματος χάρη στην Ιαπωνία βλέπουμε τεχνητή νομοσύνη σε συνδυασμό με γιατρούς οδηγεί σε καλύτερες διαγνώσεις και περισσότεροι άνθρωποι έχουν καλύτερη θεραπεία και πεθαίνουν λιγότεροι. Ε, με μεγάλη μου χαρά να ακούσω αυτά που θα πούν οι διάφορες θρησκείες και εκκλησίες επί του θέματος, αλλά αν το δούμε το θέμα ιστορικά, και εγώ μιλώ ως χριστιανός, οι θρησκείες ε, της ανθρωπότητας δεν έχουν δείξει να θέλουν να αγκαλιάσουν την τεχνολογία. Ξεκινήστε με τον Γαλιλαίο και πολύ αργότερα πολλές φορές η θρησκεία ε, δεν αγκαλιάζει την τεχνολογία για λόγους που μετά από ένα αιώνα μοιάζουν παράλογοι. Ε, γι' αυτό είμαστε στην πολιτική για να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι λογικό να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία. Πρέπει βέβαια να έχουμε ένα κώδικα ηθικής, να έχουμε ε, καλές πρακτικές και να καταδικάζουμε τις κακές, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα και αν στην Ευρώπη εφαρμόσουμε μια πολύ περιοριστική προσέγγιση, οι επενδύσεις και οι θέσεις θα πάνε κάπου και εμείς απλά θα επηρεστούμε αρνητικά αντί να επωφεληθούμε από την τεχνητή νομοσύνη. Το βλέπετε στην Ευρώπη. Πριν από 200 χρόνια οι χώρες που αγκάλιασαν την ατμομηχανή ήταν εκείνες και που προχώρησαν γρηγορότερα και χώρες όπως η Ρωσία που δεν το έκαναν έμειναν φτωχές για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε καθυστέρηση. Εγώ λοιπόν θέλω την τεχνητή νομοσύνη, θέλω κώδικα ηθικής, θέλω διαφάνεια, θέλω να εξηγούνται τα πράγματα. Και επίσης ε, θέλω να εκπαιδευτούν οι νέοι ε, να αποκτήσουν δεξιότητες, τις απαραίτητες, αλλά και πολλοί ενήλικες που ε, θα χάσουν η σωστή δουλειά τους λόγω τεχνητής νομοσύνης. Αυτό όμως δεν είναι λόγος για να μην τη στηρίζει την τεχνητή νομοσύνη. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι και να είναι πιο παραγωγικοί στο μέλλον. Ε, πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ε, ερωτήσεις λοιπόν, παρακαλώ. Βλέπω έχετε ερωτήσεις να υποβάλλετε. Ας ε, πάρουμε τις ε, πρώτες τέσσερις ερωτήσεις, γιατί δεν είμαι και σίγουρη ότι έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, ευχαριστώ. Πριν από μερικά χρόνια συμμετείχα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα συμπόσιο για τους κινδύνους ε, των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για τα κινητά τηλέφωνα. Και ανακάλυψα ότι το συμπόσιο αυτό χρηματοδοτήθηκε από τους κατασκευαστές των κινητών τηλεφώνων. Καλέσατε εμπειρογνώμονες και οι μελέτες τους αμφισβητούσαν τις αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία των ανθρώπων. Εγώ όμως ως απλός πολίτης ε, Κανείς εδώ δεν μίλησε για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Μπορεί να δημιουργήσει απασχόληση, ε, αν καν το, το εγκρίνουμε αυτά μετά τα 5G. Ε, ναι, θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης στις, ε, ε, τα νοσοκομεία, γιατροί κτλ. Εδώ όμως δεν ακούσαμε τίποτα από αυτού. Επίσης λέτε για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ναι, θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης στην Κίνα και στη Silicon Valley της Ινδίας και εδώ στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθούν τεστ και θέσει απασχόληση που θα προκύψουν δηλαδή από την ανάπτυξη τη τεχνητή νοημοσύνη. Μίλησε η κυρία προηγουμένω ε, ε, για το Ισλάμ ε, και για την θέση του Ισλάμ. Δεν είναι ερώτηση, διότι με ενδιαφέρει τόσο το θέμα αυτό που λυπάμαι που δεν ακούω του ομιλητέ να μιλάνε για αυτό που πραγματικά αγγίζει τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το δεύτερο ερώτημα, παρακαλώ. Ο κύριος εδώ, ναι. Ναι, ευχαριστώ. Το όνομά μου είναι Στίβεν Μπάλκμους. Είμαι στην ε, Μεγάλη Στοά του Βελγίου ε, και είμαι και σύμβουλος ζητήματα της νοημοσύνης και διαχείρισης και management. Ε, ε, μια από τους βασικούς πυλώνες ε, ε, της μασονίας είναι να βασιζόμαστε σε συγκεκριμένε παραδόσεις και κάτι που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτόν τον ενδιαφέρον κατάλογο των δεξιοτήτων των πολιτών είναι η καλύτερη γνώση της ανθρώπινης νοημοσύνης. Πολύ σωστά θέλουμε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να μπορούν να είναι διαφανή και εξηγήσιμα. Έχουμε όμως ποτέ σκεφτεί κατά πόσο η ανθρώπινη νοημοσύνη έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα όταν έχουμε πράγματα όπως το ένστικτο και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις όπου χρησιμοποιούμε το ένστικτό μας. Ε, στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πολύ καλά από πού προέρχεται αυτό το ένστικτο. Βεβαίως προέρχεται από πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει, από τα δικά μου δεδομέ, από τα δικά μα δεδομένα και δίκτυά μας, αλλά δεν ξέρουμε, ξεχνάμε από πού προέρχονται αυτές οι γνώσεις συχνά. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι τα παιδιά και ο κάθε πολίτης ε, ουσιαστικά να γνωρίζει ποια είναι ε, τα θετικά στοιχεία και οι αδυναμίες της ανθρώπινης νοημοσύνης. Ε, είναι οι ίδιοι οι κίνδυνοι που υπάρχουν και στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή να είναι ατελείς οι γνώσεις, να είναι μεροληπτικές, να μην υπάρχει ποικιλομορφία στον τρόπο που μαθαίνουμε κάποια πράγματα και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Νομίζω ότι ε, ο καθηγητής Μέτσιγκερ που έχει γράψει εξαιρετικά βιβλία για την ε, ε, συνείδηση μπορεί να συνεισφέρει σίγουρα προς την κατεύθυνση αυτή για το πώς δηλαδή μπορεί να υπάρχει καλύτερη κατάρτιση σε, ζητήματα, σε τέτοια ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ ο Πάτερ Γιώργος Λέκας από την Εκκλησία της Ελλάδας. η πιο μεγάλη οργάνωση ε, μη κερδοσκοπική υπέρ της, ε, ε της προόδου. Ε, ε, το 2018 σε μια έκθεση της λέει θα πρέπει τα συμβιωτικά αυτόνομα συστήματα να αναπτύσσονται με βάση τις επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Και λέμε εδώ το SAS, Symbiotic Autonomous System, μπορεί να προβλέψει τη σταδιακή συμμετοχή των σούπερ με, με μη προσδιορισμένο αριθμό ε, ε, συστατικών ε, συνισταμένων στα πλαίσια του αργορίθμου. Οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί να είναι όλο και πιο ανυπεράσπιστοι για το πώς το SAS τελικά ελέγχει όλα, όλα τα στοιχεία λήψης αποφάσεων, τα πιο σημαντικά. Μπορούμε αυτά να, γίνουν μέσω τελελογικής αυτοργάνωσης ή πρέπει να είναι αντικείμενο ε, διεθνών πολιτικών ε, αποφάσεων. Αυτό το θέμα δεν έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο κρατηρίων που συζητήθηκε σήμερα. Γνωρίζουμε το, την απάντηση αυτό χάρη ε, στην πολύ ε, ειλικρινή παρουσίαση του κ. Μέτσιγκερ. Όπω και να, έχω, να έχει κρατήσει γραμμέ όπω αυτέ που συζητούμε σήμερα, δεν μπορούμε να μα προστατεύσουν από ένα μέλλον χωρί ανθρώπου ε, που ουσιαστικά διακυβεύει τον άνθρωπο όπω το ξέρουμε σήμερα, την ύπαρξη των ανθρώπων όπω το ξέρουμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι πρέπει οπωσδήποτε ε, όταν ότι πρόκειται για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα όταν γίνονται έρευνε επιστημονικέ προ την κατεύθυνση αυτή και πρέπει να διώκονται ποινικά. Πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο τελικά είναι προτεραιότητά μα στην Ευρώπη να, ε, οι επενδύσει ή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ ακόμα μία κυρία έχει το λόγο. Uh, um, There was a high level group on disinformation. Να ρωτήσω κάτι από τις γραμμές. Ετοιμάστηκε ένα πολύ καλό έγγραφο σε ό,τι αφορά την, παραπληροφόρηση και τελικά είχαμε ένα θελοντικό κώδικα για την παραπληροφόρηση και τις διάφορες πλατφόρμες. Ε, και πήραν αυτό τη θελοντική δέσμευση να σεβαστούν αυτόν τον κώδικα οι μεγάλες πλατφόρμες με ετήσιες ε, ε, εκθέσεις για την πρόοδο. Είμαστε δύο μήνες πριν τις εκλογές τώρα και το Facebook, ε, το Twitter, η Google δεν, έχουν, δεν παίρνουν διαφανείς αποφάσεις ούτε για τις διαφημίσεις, ούτε για τους αλγόριθμους. Ουσιαστικά δηλαδή δεν κάνουν κάτι. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί. Γίνεται μια πολύ ωραία δουλειά στην ομάδα υψηλού επίπεδου, που οδηγεί σε υπέροχε κατευθυντήριε γραμμέ και τελικά η Κομισιόν λέει εντάξει, αυτό εθελοντικό, εθελοντικά όμω. Ε, έχουμε κώδικα καλή πρακτική για τι πλατφόρμε ε, και τελειώσαμε με την ηθική τη τεχνητή νοημοσύνη. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτό που έκανε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή να έχουμε κάτι ισχυρό, κάτι υποχρεωτικό διότι συνεδριάζουν ε, οι εμπειρογνώμονε, γίνεται πολύ καλή δουλειά, η Κομισιόν συμφωνεί και τελικά δεν οδηγούμαστε σε κάποιο απτό αποτέλεσμα. Α εξασφαλίσουμε λοιπόν αυτή τη φορά θα υπάρχει μια νομοθεσία δεσμευτική. Ναι, ένα ερώτημα ακόμα εκεί πίσω. Δυστυχώ ε, δεν υπάρχει χρόνο για κάποιον άλλον. Um, Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι, ε, ασκούμε στο ερευνητικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και γράφω και εγώ την διατριβή μου για, την, ε, για τα θέματα που συζητάμε. Η δική μου προσέγγιση προς την τεχνητή νομοσύνη, η στάση μου είναι ότι φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Η σχέση μου έχει σχέση και με αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αφενός ένα περιβάλλον φιλικό προς επιχειρήσεις και αφετέρου προστασία των πολιτών από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ε, γνωρίζουμε λοιπόν και δεχόμαστε ότι είμαστε δύο βήματα πιο πίσω στο να εντοπίσουμε το περιεχόμενο, ε, την προέλευση του περιεχομένου, των αλγορίθμων, ε, τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και ρωτώ, αν δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την ε, πηγή, τότε ποια είναι η εναλλακτική λύση για τις πλατφόρμες, αυτές είναι υπεύθυνε και οι host και το δεύτερο κομμάτι της ερώτησής μου είναι ως εκπρόσωποι των πολιτών έχουμε την υποχρέωση να προστατεύουμε τους πολίτες και πώς δικαιολογούμε ότι δεν ε, προτιμάμε το δεύτερο ε, νομοθετικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. Ε, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο σε όλους ε, τους ομιλητές ε, για να κάνουν κάποια σχόλια και να δώσουν κάποιες απαντήσεις, διότι θίγησαν σημαντικά θέματα. Παρακαλώ, κύριε Μέτσιγκερ. Πρώτα απ' όλα, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Η τελευταία εκδοχή αυτών των κατευθυντήων γραμμών ηθικής ε, που θα δείτε είναι πολύ καλύτερες από το σχέδιο που είδατε το Δεκέμβρη και θα είναι και πολύ καλύτερο από οτιδήποτε έχουν η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα είναι κάτι πραγματικά σημαντικό. Εγώ είμαι καθηγητής ε, φιλοσοφίας. Έχω πολλά προβλήματα ε, σπάζω κεφαλιά, δεν είμαι ικανοποιημένο με το τελικό ε, κείμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καλύτερο από ό,τι υπήρχε μέχρι σήμερα. Αυτό που έμαθα τους τελευταίους εννέα μήνες είναι να υπάρχει ε, νομοθεσία που να μπορεί να εφαρμόζεται και είχα πραγματικά πολύ περισσυζητήσει με εκπροσώπους του νομικού κόσμου που μου είπαν ότι για εννέα χρόνια υπήρχαν κάποιες προσπάθειες και υπάρχει αυτό που εμπειρογνώμονες αποκαλούν ε, ως ε, μια εξέλιξη που είναι πολύ πιο γρήγορη από ό,τι μπορούν να ανταποκριθούν οι δημοκρατικοί ε, θεσμοί. Ίσως πρέπει να επενδύσουμε και σε νέα μοντέλα διακυβέρνησης, έτσι ώστε τα κενά στον βηματισμό, όπως λέγονται, να είναι μικρότερα και να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Θα ήθελα να απαντήσω σε μία από τις ερωτήσεις που ετέθησαν από το πίσω μέρος της αίθουσας. Στην παρούσα κατάσταση δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, δεν μπορούν ε, να είναι υπόλογες οι πλατφόρμες, αλλά αυτό πρέπει να το επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα οδήγησε την Google και άλλους εκτός της χώρας. Είναι και αυτό μια επιλογή. Εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε την επιλογή ε, το Facebook να μην λειτουργεί στην Ευρώπη αν τα πράγματα γίνουν ανεξέλεγκτα, παραδείγματο χάρη στις επόμενες εκλογές. Εγώ δεν στηρίζω κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση για να ε, αναλάβουν οι μεγάλοι πάροχοι τις ευθύνες τους. Αλλά δεν ήθελα να αφαιρέσω άλλο χρόνο από τους ε, συναντέλφου μου. Θέλει κάποιος να σχολιάσει. Από ό,τι βλέπω όχι. Πολύ ωραία. Ashley θέλετε εσείς ε, να έχετε την τελική λέξη. Ίσως ε, να απευθυνθώ στην κυρία που έκανε την ερώτηση από το πίσω μέρος της αίθουσας και είπε ότι φοβάται πάρα πολύ. Εγώ σας λέω να μην φοβάστε, να είσαστε αισιόδοξοι. Η ζωή βελτιώνεται. Ε, σήμερα στον κόσμο έχουμε πολύ λιγότερους που πεινάνε από ό,τι υπήρχαν κατά το παρελθόν. Η, ε, ο κόσμος προοδεύει, η τεχνολογία μας κάνει πιο πλούσιους, Σήμερα, όπως σας είπα, θα πεινάσουν πολύ λιγότεροι από ό,τι πίναγαν πριν από 10-20 χρόνια. Βεβαίως, η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι καλό ή κάτι κακό. Αυτό ισχύει και με το διαδίκτυο, το βλέπω και με τα παιδιά μου. Ε, δεν μπορεί κανείς να σταματήσει την ε, τεχνητή νοημοσύνη, απλά να τη χρησιμοποιεί σωστά, να πει στους νέους ανθρώπους ότι τα μέσα κοινωνικής βελτίωσης ε, είναι χρήσιμα, αλλά αν περνάει κανείς κάθε μέρα 8 ώρες πάνω σε αυτά, μπορεί να βλάψουν τη ζωή τους. Ε, διασπορά ψευδών ειδήσεων, πάντα υπήρχαν αυτά. Πίσω από 100 χρόνια και όλοι καταδικάζουν ε, τη Βρετανική Αυτοκρατορία ότι ήταν αυτή ε, που έλεγε πάντα ψέματα και έσπηρε φήμες. Αλλά να σας πω κάτι. Η προπαγάνδα και οι ψεύτικες ε, ειδήσει, οι φήμες υπάρχουν από τότε που υπάρχει ανθρωπότητα. Μόνο οι πλατφόρμες άλλαξαν. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε αισιόδοξοι, ας είμαστε θετικοί, ας αγκαλιάσουμε αυτήν την τεχνολογία που θα βελτιώσει τη ζωή όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ και με αυτή την αισιόδοξη κατακλίδα να κάνω εγώ ε, μια σύντομη παρατήρηση και να δώσω το λόγο στην κυρία Αντιπρόεδρο. Να πω ότι επειδή έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ε, τα deepfakes ε, θα συμπεριλαμβάνουμε και αν εντοπίζει κάποιος από εσά μία πραγματικά ψευδή είδηση, πρέπει να την αναδεικνύει. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει για να εντοπίσουμε αυτά τα ψεύδη και τις ψευδείς ειδήσει. Δεν χρειαζόμαστε ε, ε, ειδικό ε, τομέα που να ασχολείται με την αλήθεια ή όχι. Ε, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες και να τους δώσουμε περισσότερες αναλλακτικές λύσεις για το πώς αναζητούν ε, και χρησιμοποιούν τα δεδομένα. Κατάλαβα ότι αν συμφωνήσουμε πάνω στις ανθρώπινες αξίες ε, και νομίζω όλοι συμφωνούν ε, με τις ανθρώπινες αξίες, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με σωστό και κατάλληλο τρόπο, ας πούμε, για να ε, προβλέψουμε ασθένειες. Αλλά εμείς θέλουμε να στηρίξουμε την καλή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτό. Δεν είναι το τελικό σχέδιο, είναι ένα σχέδιο που είναι δυναμικό, ε, που ε, μας ε, κρατάει σε επαφή με την τεχνολογία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε φιλικοί προς τις καινοτομίες και να μην τις αναχαιτίζουμε λόγω φόβου. Θα δώσω βέβαια το λόγο στην κυρία Μαγκίνες για τις τελικές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το θαυμάσιο διάλογο και νομίζω ότι αυτή είναι απλά η αρχή. Ευχαριστώ κυρία Καηλή.